τέλος της συνόδου θα εγκριθούν αυτές οι ε, υποψηφιότητες. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι δυνάμει του άρθρου 74 του κανονισμού του Κοινοβουλίου μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, συνυπέγραψα έξι νομοθετικές πράξεις υπό την τακτική νομοθετική διαδικασία οι οποίες θα δημοσιευθούν στα πρακτικά του ε, Κοινοβουλίου της τρέχουσας συνόδου και πιστεύω ότι ο κύριος Κονπεντήτ θα αισθανθεί ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ε, έγκριση των πρακτικών αυτών και σημειώνω παρακαλώ στα πρακτικά τον, ε, ε, τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του κυρίου Κόνβεντιτ. Επίσης κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης